Då eh, όλοι. Θέλω να αρχίσουμε. Ε, σας καλωσορίζω μετά τις ε, καλοκαιρινές ε, διακοπές. Κάναμε σύσκεψη με τους συντενιστές νωρίτερα. Το σημείο δίνει είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει καμία πρόταση. Ε, τροποποίησης, οπότε θα θεωρούμε εγκεκριμένα. Κατόπιν σημείο 3 ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω το Χαρινάκη Σαβαλμπέιτα Φερνάντες από την Ισπανία, νέο μέλος. Καλωσορίσατε. Και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι την επόμενη συνεδρία θα την κάνουμε στο Στρασβούργο. Ή μάλλον μία επόμενη συνεδρίαση, όχι η μαλλον μια επομενη στο Στρασμούργο. οχι η επομενη θα γίνει ε, στις 7, ε, ε, στις 20, την 21η Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Αλλά δεν είναι η επόμενη, είναι η μεθ επόμενη και ούτω ή άλλω συνεδριάζουμε και το Σεπτέμβριο. Αλλά ήθελα να σα πω ότι η συνεδρία του Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο. Ε, στις 10 Ιουλίου ε, έγινε και συνεδρία των συντονιστών. Σα έχουμε στείλει τα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. μπορούμε να εγκρίνουμε όλα τα πρακτικά όπω προβλέπετε στο σημείο 5. 4. Στη συνέχεια έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 21 και 22 Νοεμβρίου 2011, 9 Φεβρουαρίου 2012, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2012 και 21 Μαρτίου 2012. Αυτά. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Τρεις εκθέσεις έχουμε και θα μιλήσω στα αγγλικά. Ε, θα αρχίσουμε τις ε, ψηφοφορίες μας. Επαναβιομηχανιοποίηση της Ευρώπης για την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας και της αηφορίας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Παπαδοπούλου αν θέλει το λόγο. Θα το αρχίσουμε. Όχι. Ωραία, ας αρχίσουμε τότε. Α, επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι δύο εξημών και ο υποφαινόμενος σε αυτούς τους δύο ξέχασαν τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Ε, αν χρειαστεί θα προσθέσουμε τις ψήφους. Ας αρχίσουμε με την πρώτη τροπολογία. Παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Ναι, και εγώ, και εγώ ξέχασα την κάρτα μου, ζητώ συγγνώμη. Ε, είναι που ήταν οι καλοκαιρινές διακοπές και νιώθαμε όλοι ελεύθεροι και αυτά δεν πειράζει. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Επαλήθευση. Τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την τροπολογία 7 παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 8 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε στη 14 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 13 και 15 καταπίπτουν, 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά, αποχές Πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε. Ποιοι είναι υπέρ της 17 κατά αποχές. Αγκρίθηκε. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Για το σύνολο της ε, γνωμοδότησης παρακαλώ. Παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Ξεκάθαρα εγκρίθηκε ομόφωνα. Περνούμε στο σημείο 7, δηλαδή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις Αχέλ, συμβαστική 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 τώρα που είναι κατά τμήματα, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15 έχει αποσυρθεί. 16 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 17. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Η 18 καταπίπτει, 19 τώρα. Υπέρ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 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 41 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44. Κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο σημείο 8. Γενικός προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014. Όλα τα τμήματα. Δεν είναι εδώ η συγγήτρια, λέμε πως είναι κάποιος άλλος εδώ που θέλει να πάρει το λόγο εκ μέρους της συγγήτριας. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε ψηφίζουμε. Και αρχίζουμε με την τροπολογία 6240. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6203. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 62-19. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 62-18 τώρα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 62-17. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 62-06. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62, 22 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 62, 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62, 31 και 62-12 καταπίπτουν. 62-13 τώρα λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-51 υπέρ, κατά, αποχές, η τελευταία είναι μια προφορική τροπολογία, οπότε πρέπει να ρωτήσω πρώτα αν υπάρχει αντίρρηση να υποβληθεί σε ψηφοφορία η προφορική. Πρόκειται για την 6253. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία. Ας ψηφίσουμε τότε την τροπολογία. Προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε το σύνολο. Άρα έληξε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, θα επιστρέψω στα Σουηδικά, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες, θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Στο σημείο 9 θα περάσουμε γυναίκες με αναπηρία. Η συγγήτρια, η κυρία Βέρτμαν, θα πάρει πρώτο λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τον λόγο, Πρόεδρε. Έχουμε 196 τροπολογίες και νομίζω πως ε, κάθε ένας από τους συναδέλφους μου αξίζει ευχαριστειών για την πρωτοβουλία και την δουλειά που έκαναν. Προσπαθούμε να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες, συνεχίζεται ακόμα η προσπάθεια. Έχουμε κάποιους πολύ καλούς συμβιβασμούς. Πιστεύω πως πολλές τροπολογίες ήταν χρήσιμες, αρκετές ήταν αρκετά μακροσκελείς. Εξαιρέσεις βέβαια ήταν αυτές, ορισμένες άλλες τροπολογίες ε, επαναλαμβάνονται, είναι παρόμοιες. Προς το παρόν το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς και θα ενημερώσουμε τους κοιόδης εισηγητές αυτό το χρόνο έτσι ώστε να λάβουμε την σύμφωνη γνώμη τους και θα επιστρέψουμε το στομότερο δυνατόν με την ψηφοφορία. Να σας ενημερώσω επίσης ότι υπάρχει μία τροπολογία, η τροπολογία 1, η οποία, να σας ενημερώσω ότι εφο, εάν εγκριθεί, θα αναβληθούν τα πάντα. Θα πρέπει να ζητήσουμε εκ νέου υποβολή έκθεσης με νέο τίτλο και στην περίπτωση αυτή δεν γνωρίζουμε πότε θα πάει η έκθεση στην Ολομέλεια. Είναι μια αναβολή δηλαδή για χάρη αναβολής. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, Πρόεδρε, η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει γίνει πολλή δουλειά από πολλούς συναδέλφους και δεν πιστεύω ότι πρέπει να καθυστερήσουμε περισσότερο. Απλά να σας επιστήσω την προσοχή λοιπόν σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, θα καλωσορίσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Mrs. please. Κυρία Παπαδοπούλου. Chair. Πρόεδρε, είμαι σκιώδης η συγγήτρια για τους σοσιαλιστές θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι η έκθεση αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τις σχέσεις, την εμιτρότητα, την οικογένεια, την οικογενειακή ζωή, σεξουαλικότητα, προστασία από την βία και από την κακοποίηση, προστασία των γυναικών που είναι θύματα κακοποίησης ή διακρίσεων εξαιτίας της αναπηρίας τους, και επειδή είναι γυναίκες και επειδή έχουν αναπηρία. Πιστεύω ότι 196 τροπολογίες που έχουμε στοχεύουν στη βελτίωση της έκθεσης. Όλοι στοχεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, πώς δηλαδή να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, πώς να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές να έχουν μια φυσιολογική ζωή και πώς να τις βοηθήσουμε να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες στην κοινωνία μας. Στηρίζω λοιπόν απόλυτα την γνωμοδότηση της κυρίας Βέρτμαν και συμμερίζομαι την άποψή της ότι θα μας δημιουργούσε πρόβλημα εάν αναβάλαμε την ψηφοφορία. Πιστεύω πως η έκθεση ως έχει είναι ικανοποιητική. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Έχουμε καταβάλει όλες οι πολιτικές ομάδες μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε την έκθεση και πιστεύω πως θα είναι το καλύτερο για όλους αν ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Η έκθεσή της είναι πράγματι μια αναγκαία έκθεση και το περιεχόμενό της είναι σημαντικό. Εμείς υποβάλαμε εκ μέρους του ΕΛΚ 40 κάτι τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο να βαθύνουν ακόμα περισσότερο σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες με αναπηρίες, ιδιαίτερα τα θέματα προσβασιμότητάς τους. Βλέπετε, στην Επιτροπή ετοιμάζουν ένα νόμο για την πρόσβαση ακριβώς των ατόμων αυτών, θα προχωρήσει φέτος και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι βέβαια μόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλες τις ε, περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ε, ζωή ενός ατόμου με αναπηρία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η προσβασιμότητα πρέπει να είναι πλήρης. Δεν έχει να κάνει μόνο με την αρχιτεκτονική των κτηρίων, έχει να κάνει όμως και με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής των γυναικών αυτών. Είτε πρόκειται για την εκπαίδευση που να μπορούν να συμμετέχουν, είτε πρόκειται για την υγεία που να δεν συμπεριλαμβάνει και αυτές, είτε οτιδήποτε άλλο στην κοινωνία μας. Στην Επιτροπή εγκρίθηκε μία οδηγία για τα ψηφιακά ζητήματα. Μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες τα ψηφιακά περιεχόμενα, γι' αυτό και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι γυναίκες με αναπηρία. Να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε να μπορούν να αποφεληθούν από το διαδίκτυο και τα άτομα με αναπηρία εκείνα τα οποία δεν βλέπουν αρκετά καλά το οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τις γυναίκες αυτές. Επίσης υπάρχει μια τροπολογία για την κατάρτιση στον τομέα της υγείας και στην εκπαίδευση προκειμένου να μπορούν και τα άτομα αυτά να συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Υπάρχει επίσης και ένα τμήμα το οποίο αφιερώνεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα αντισυλληπτικά. Πρέπει να υπάρχει συνένεση από τη γυναίκα με αναπηρία για να πάρει αντισυλληπτικά. Διότι πολλές γυναίκες με αναπηρίες θέλουν να κάνουν παιδιά. Υπάρχουν επίσης και ένα που αναφέρονται στην αγορά εργασίας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στα επίπεδα που προτείνουμε με τη στρατηγική 2020 για την ένταξη στην αγορά εργασίας, αυτό δεν θα επιτευχθεί αν δεν συμπεριλάβουμε στην αγορά εργασίας και τις γυναίκες με αναπηρίες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας των ε, γυναικών με αναπηρίες. Δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνονται οι προσαρμογές που πρέπει στους χώρους εργασίας για να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι γυναίκες με αναπηρίες. Έχουμε και μία τροπολογία που ζητά από τα κράτη-μέρη να συμπεριλάβουν δείκτες για τις γυναίκες με αναπηρίες ώστε όταν εξετάζονται τα διάφορα θέματα να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών με αναπηρία στην κάθε περίπτωση. Και έτσι να αντιληφθούμε καλύτερα ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας με αναπηρίες είτε στις εθνικές αγορές είτε στην ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα. Και ζητάμε επίσης από τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στατιστικές και στοιχεία που να αναφέρονται στη σχέση των δύο φύλων για να δούμε κατά πόσο υπάρχει κάποια διάκριση σε βάρος των ε, γυναικών. Η βία, η ενδοοικογενειακή, όντως είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που έχουμε γυναίκες με αναπηρία. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μέτρα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστούμε κυρία Τσούμπε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ε, συμφωνούμε εν γέννη ως προς τη βάση της πρότασης ε, που κατέθεσε η συγγήτρια. Προτείναμε κάποιες τραπολογίες που ως πλήστον αποσκοπούν στο να επιστήσουν την προσοχή στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες με αναπηρία όχι μόνο διότι είναι γυναίκες και επειδή έχουν αυτή την αναπηρία, αλλά ε, οι γυναίκες που ζουν σε χώρες όπου τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα με αναπηρίες ε, παρουσιάζουν ατέλειες, ε, γίνονται θύματα τέτοιων διακρίσεων. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την προώθηση των δυνατοτήτων τους και αυτό είναι συνάρτηση του κοινωνικού στρώματος στο οποίο ανήκουν. Είναι απαραίτητο ως εκ τούτου να αυξηθούν οι επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας δεν είναι αυτό το αντικείμενο όλων των τροπολογιών, αλλά ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως ως προς τις υπηρεσίες για τη σεξουαλική, σεξουαλική συγγνώμη, και αναπαραγωγική υγεία ε, για τα άτομα με αναπηρίες ε, ε, καθιστά απαραίτητη παρουσία εξειδικευμένων επαγγελματιών του κλάδου υγείας, κυρίως σε περιπτώσεις επιπλοκών της εκκίνησης, της εγκυμοσύνης, Επίσης τονίζουμε ότι ιδιαίτερα είναι τα προβλήματα όταν είναι διανοητική η καθυστέρηση, υπάρχει κάποια άλλη διανοητική αναπηρία. Αυτά τα μέτρα λιτότητας, όπως αποκαλούνται, η περικοπή των δημοσίων δαπανών, που δεν είναι δαπάνες, επενδύσεις είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτά τα μέτρα αυξάνεται, μάλλον επιδεινώνεται η κατάσταση αυτών των γυναικών, περιορίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες, στην κατάρτιση, στον αριθμό των θέσεων για τους επαγγελματίες στον τομέα υγείας που είναι οι μόνοι που μπορούν να ασχοληθούν με τέτοιες γυναίκες διότι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και πολλές φορές υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις για αυτές τις θέσεις ε, περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση, περιορισμός της ε, κατάρτισης των ε, ειδικευμένων επαγγελματιών ε, που θα συνοδεύσουν αυτές τις γυναίκες τόσο για την κατάρτιση όσο και για την απασχόληση αυτών των γυναικών. Θα πρέπει να αναστραφεί λοιπόν αυτή η τάση Ε, και να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός που είναι απόρρια αυτών των μέτρων. Στη συνέχεια, σε άλλες τροπολογίες, τονίζουμε πόσο μεγάλες ε, είναι οι δυνατότητες, πόσο μεγάλη είναι η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει ο κάθε ένας από εμά στο σχολείο, στη δουλειά, όπου βρίσκεται. Θα πρέπει να τονιστεί και αυτή η συνιστόσα. Όχι μόνο όμως, να τονιστεί και η σημασία της οικογένειας και ε, τα άτομα με αναπηρίες ε, όταν διαβιούν στους κόλπους της οικογένειάς τους ε, έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Εξάλλου, ως προς τις κρατικές δαπάνες είναι και η φθηνότερη λύση. Τονίζουμε επίσης τροπολογίες, ε, κάτι που κρίνουμε σημαντικό χάρη στα δεδομένα που συλλέξαμε. Με την αύξηση της φτώχειας είναι ανησυχητικό ότι αυξάνεται και η σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών με αναπηρίες. Είναι ένα τραγικό φαινόμενο που θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να καταπολεμηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Τζάστε, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μοχσέ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια και τα μέλη του Κοινοβουλίου για όλες τις τροπολογίες. Όπως προαναφέρθηκε, οι μη διακρίσεις και η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020. Συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου σε όλε τι επιτυχίε τη στρατηγική και επίση και συμπεριλαμβάνεται σε δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση της οικονομικής ανεξαρτησίας Προσπαθούμε λοιπόν εκεί να συμπεριλάβουμε την ε, διαστάση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, στην έκθεση Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αναπηρίας, η οποία θα δημοσιευθεί μέσα στο 2013, συμπεριλαμβάνονται αυτές οι προτάσεις. Επίσης, να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν αναφερθεί ως πιθανός ε, Στόχο μία μιας πρόταση, η οποία άρχισε τον Μάρτιο του 2013 για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των κρατών μελών για τα άτομα με αναπηρία. Και επίσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας στις πιο ευάλωτες ομάδες, για παράδειγμα τις γυναίκες με αναπηρία. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν επίσης την δυνατότητα να αναπτύξουν προγράμματα καταπολέμησης των ανισοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Βέρτμαν ε, για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρεμβάσεις και τις τροπολογίες τους. Όπως αναφέρα και στην αρχή, προσπαθήσουμε να συλλέξουμε όλες τις απόψεις των γρηγορότερο δυνατόν και να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στις 3 Οκτωβρίου εδώ στην Επιτροπή και το Νοέμβριο θα περάσει ε, από την Ολομέλεια η έκθεση 23 και ολοκληρώνουμε τώρα το σημείο ε, ναι, Θα περάσουμε στο σημείο 10. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα. Η αντιπρόεδρό μα η συγγήτρια, η κυρία Εστρέλα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή σας, για καταθέσατε 217 τροπολογίες. Αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Πραγματευόμαστε ε, και ως επιτοπλίστων συμφωνώ με μεγάλο αριθμό αυτών των τροπολογιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες, ε, Γκαμπριέλ, Μογάν Σαχτιέ, Ματέρα, ε, Γκαρσία Πέρες, ε, Ζήτα Μπουρμάη, ε, Σοφία Ιντβελντ, ε, η κυρία Κορνέλισεν, ο κύριος Γκούσταυσον, η κυρία Τσούμπερ και άλλοι, για να τους απαριθμίσω όλους, κατέθεσαν τροπολογίες που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχομένου της έκθεσής μας. Όμως, Υπάρχουν και κάποιες που δεν μπορώ να αποδεχθώ, διότι αμφισβητούν αρχές και κεκτημένα δικαιώματα καθώς και συμβαστικές λύσεις, οποίες έχουμε καταλήξει σε διεθνές επίπεδο, κατόπιν διαβουλεύσεων ε, από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναλυθεί ε, και να εγγραφεί στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πέραν αυτού είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε την ισότητα των δύο φύλων. Υπάρχουν τροπολογίες που προτείνουν να νερεθεί ισχύουσα νομοθεσία κυρίως σε σχέση με το θέμα της έκτρωσης. 20 κράτη-μέλη, υπενθυμίζω, ε, αναγνωρίζουν ως νόμιμη την έκτρωση. Από τους υπόλοιπους, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κύπρος και η Φινλανδία ε, επιτρέπουν μια ευρία ερμηνεία των εφιστάμενων περιορισμών και τώρα ε, το, η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Μάλτα έχουν πιο περιοριστική ερμηνεία. Ε, και στη Μάλτα μάλιστα δεν υπάρχουν και νομικές εξαιρέσεις. Ε, απαγορεύεται η έκτρωση δια νόμου. Πολλές ε, γυναίκες ταξιδεύουν σε άλλα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μπορέσουν να διακόψουν εκεί την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη τους. Αυτή η απαγόρευση που ισχύει σε διάφορα κράτη-μέλη πλήττει περισσότερο ε, τις γυναίκες ε, που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, δεν έχουν ίσως την ε, απαιτούμενη εκπαίδευση, δεν έχουν τους πόρους για να ταξιδέψουν με ευκολία σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν έτσι πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτρωσης δεν έχουν ίσως την κατάλληλη κατάρτιση, ενημέρωση ή οικονομικούς πόρους, δεν έχουν σε κάθε περίπτωση τις ίδιες δυνατότητες ε, να προσφύγουν ε, σε υπηρεσίες άλλων κρατών. Λόγω αυτού ε, διωγγώνεται η ανισότητα που διαπιστώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας το κόστος ε, μιας ασφαλούς έκτρωσης ε, αντιστοιχεί στο 1 δέκατο του κόστους της περίθαλψης ε, λόγω επιπλοκών, λόγω μη ασφαλούς έκτρωσης. Υπάρχουν βεβαίως και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ε, ε, ψυχικά προβλήματα, συναισθηματικά προβλήματα και ούτω καθεξής, πέρα από αυτό το κόστος που υπολογίζεται δηλαδή. Σε άλλες τροπολογίες ε, διαπιστώνω ότι επαναλαμβάνουμε το ίδιο περιεχόμενο Και έχω την εντύπωση ότι έρχονται αυτέ οι τροπολογίε από άλλου διεθνεί οργανισμού εκτό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι βουλευτέ απλώ τι κατέθεσαν επαναλαμβάνοντα το περιεχόμενο τη έκθεσή μου. Στη συνέχεια υπάρχει το θέμα τη αντίρρηση συνείδηση, συλλογική και όχι μόνο ατομική. Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιε τροπολογίε. Καθώ επίση και τροπολογίε που θέτουν να αμφιβόλω και το θέμα της σεξουαλικής αγωγής των παιδιών και των εφήβων. Εδώ τίθεται ζήτημα ισότητας των δύο φίλων Αυτές οι τροπολογίες που ε, αμφισβητούν αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης στη σεξουαλική αγωγή είναι απαράδεικτες ε, κατ' εμέ. Κατόπιν, Υπάρχουν άλλες ε, τροπολογίες ε, που σχετίζονται με τον ορισμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων. Μα αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτόν τον τίτλο και δεν πρόκειται να προσφύγουμε σε άλλες, ε, σε αναδιατύπωση του ορισμού και του τίτλου. Κατόπιν άλλες τροπολογίες που αμφισβητούν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της υγείας και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και υγείας στα κράτη-μέλη οφείλουν να συμβάλλουν ούτως ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος ε, για την επίτευξη του ε, στόχου μόνο 5 των στόχων της ε, χιλιετίας που καλύπτει την σεξουαλική υγεία, αναπαραγωγική υγεία, την υγεία των νεογνών, την, τα θέματα της μητρικής θνησιμότητας, του προγενετικού ελέγχου, την με ευτική και γυναικολογική περίθαλψη, τη προσφορά υπηρεσιών μετά τον τοκετό, ε, την ε, αντιμετώπιση σεξουαλικώς μεταδεδομένων λοιμόξεων, και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι ήδη έχουμε μία πάρα πολύ καλή βάση όπου θα εδραστούν οι συμβαστικές μας ε, τροπολογίες. Έχει προβλεφθεί σύσκεψη των σκιωδών την επόμενη Τετάρτη. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική η ευκαιρία να συναντηθούμε, να αποπειραθούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, λύσεις που θα κατοχυρώσουν την ε, απαιτούμενη ευρεία υποστήριξη όλων ε, για την πρόθεση της έκθεσης. Όλοι όσοι θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μου γνωρίζουν ήδη ότι καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι ικανοποιητική η έκθεση να ε, εγκριθεί από την Επιτροπή μας και κατόπιν από την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα αρχίσει η συζήτηση η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που τα θέματα υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας επαναλαμβάνονται στις εκθέσεις μας, δεν συνηθίζεται να έχουμε ολόκληρη έκθεση αφιερωμένη σε αυτό το θέμα. Οπότε, μπράβο, συγχαίρω την εισηγήτρια για το θάρρος της να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα που είναι περίπλοκα, που είναι ευαίσθητα και τη συγχαίρω και για το επικοδομητικό της πνεύμα διαλόγου μαζί μας από την αρχή. Θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και η συγγήτρια, αυτό με το οποίο ασχοληθήκαμε εγώ και η συνάδελφος που είναι οι νέοι. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε το θέμα των νέων και την ανάγκη να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη και την συναισθηματική οριμότητα των νέων. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτική σημασίας γιατί σήμερα ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με στερεότυπα, έρχονται αντιμέτωποι πολλές φορές με τη βία, όπου δεν υπάρχει πάντα επαρκώς ε, παρόν ο σεβασμός για τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι χρειάζεται αυτή η ίδια παιδαγώγηση γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική του υγεία. Έπειτα, μέσω της σεξουαλική και συναισθηματικής αγωγής μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους στην ζωή τους, αλλά μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε και τους γονείς και τους ενήλικες οι οποίοι συνδράμουν στην αγωγή των ε, νέων που πολλές φορές προσφεύγουν στην πορνογραφία και μπορούν έτσι να τους προστατεύσουν καλύτερα και από σεξουαλικά μεταδόμενες λοιμώξεις. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και σε μια άλλη προβληματική που επίσης είναι πολύ παρούσα στην έκθεση. Η υγεία είναι με αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει αν μη τι άλλο να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις βέλτιστες πρακτικές, να υπάρχει μια ισορροπημένη πολιτική για τα θέματα αυτά. Ο τουρισμός υγείας δεν είναι η καλύτερη λύση. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας και στο θέμα της υγείας των λεχόνων και των νεογέννητων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το θέμα της ε, εθνισιμότητας των λεχόνων. Σε πολλές χώρες μέλη, δυστυχώς, υπάρχει ως πρόβλημα και πρέπει να ανησυχήσουμε γιατί βλέπουμε μια επιστροφή προς τα πίσω σε ορισμένες χώρες παρά τις πρόοδους που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει και μια τάση να μειώνεται η παραμονή στο μευτήριο των ε, γυναικών ε, που γεννούν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Αναφέρονται στην έκθεση. Εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή Χαίρομαι που οι σκιώδεις εισηγητές θα συναντηθούν μεταξύ τους και με την εισηγήτρια και πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να πετύχουμε ένα συμβασμό για να εγκρίνουμε μια έκθεση η οποία τελικά θα είναι ισορροπημένη, θετική για τους πολίτες, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες, όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τους λιγότερο νέους και όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προβληματική αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσω εγώ με την ιδιότητα του σχεδόν εισηγητούς για αυτή την έκθεση, εφόσον δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ε, με πρόλαβε η κυρία Γκαμπριέλ. Σπάνια μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματευτούμε ένα τέτοιο ζήτημα. Συχνά απαντάτε αυτό το ζήτημα στις εκθέσεις, νομοδοτήσεις, στα ψηφίσματα, αλλά ποτέ δεν είναι το αντικείμενο της έκθεσης. Ε, είναι σπάνιο και πολύ ωραίο αυτό. Πριν το καλοκαίρι όταν έκανε την παρουσίαση η κυρία Εστρέλα πιστεύαμε και το είπαμε εξάλλου κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ότι καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων και εντάξει, ξέρουμε ότι έχετε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων και edit. Ξέρω ότι πιέστηκε, θεώρησες ότι δεν ήσουν ελεύθερη να εκφραστείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε κάποιος να πει, να σκεφτεί, να προσθέσει για αυτό το θέμα και είναι ε, ε, ε, πάρα πολύ μεγάλο και το ενδιαφέρον. Είδαμε ότι είναι πάνω από 200 τροπολογίες πιστεύω ότι υπάρχει, διαφαίνεται μια κοινή γραμμή και είπαμε ότι το θέμα είναι σημαντικό διότι σχετίζεται με τα θαμελιώδη δικαιώματα και την σεξουαλική αυτοδιάθεση των ε, γυναικών. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που συμφωνείς την πλειοψηφία των τροπολογιών που έχουν καταθέσει τα μέλη. Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι εξαιρετική σε ποιότητα η έκθεση, διότι θα, το έρισμα από το οποίο θα οικοδομηθεί το τελικό ψήφισμα είναι πάρα πολύ καλό. Χάρη στην κυρία Εστρέλα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που εργαστήκατε εξαιρετικά και μας προσφέρατε αυτή την πάρα πολύ καλή βάση για να επεξεργαστούμε τις τροπολογίες στη συνέχεια και να καταλήξουμε στην τελική έκθεση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Συνήθως ε, δίνουμε το λόγο μόνο σε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ίδια όμως η Επιτροπή ζήτησε... Ε, α, άλλαξαν τη γνώμη τους. Ε, <laughs> άλλαξαν γνώμη στο μεταξύ, ένας θα μιλήσει. Τέλο πάντων, άμα θέλετε να μιλήσετε κι άλλοι, πέρα του ενό δηλαδή, ε, έχετε το ελεύθερο από μένα, παρακαλώ. Ε, Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιο θα ηγηθεί τη έκθεση αυτή. δούμε συγγνώμη. Θα αποφασίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Συνεπώς δεν έχει οριστεί ακόμα αρμόδιος και έτσι δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να πάρουμε το λόγο. Okay, Mm, Αφού είναι έτσι τα πράγματα, θα ε, ακούσουμε και πάλι την εισηγήτρια για τις τελικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαμπριέλ που με ενθαρρύνει και σας Πρόεδρε. Και να επαναλάβω τονίζοντας ε, τη δέσμευση και την αφοσίωσή μου για την εξέβρεση συνενετικών λύσεων που θα αξίζουν την ε, στήριξη της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Γυναικών αλλά και των βουλευτών του Κοινοβουλίου όταν ψηφιστεί η έκθεση στην Ολομέλεια. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Εξάλλου, στην αρχική μου παρέμβαση ε, σας ανέφερα και εγώ, διότι καταθέσατε τροπολογίες, χάρη στις οποίες εμπλουτίζεται και βελτιώνεται η έκθεσή μου. Κρίνω λοιπόν ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ε, στο μέτρο που είναι ενδιαφέρουσε τροπολογίε όλων των πολιτικών ομάδων. Δημιουργούνται λοιπόν οι προποθέσει ε, για να καταλήξουμε ε, σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ή τουλάχιστον το ελπίζω. Ένα, μια τελική παρατήρηση και με αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι. Λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρήκε το χρόνο να διορίσει έναν αρμόδιο για αυτό το ζήτημα και δεν έχει να πει τίποτα, ε, όπως μας είπε προς το παρόν, για το ένα τόσο περίπλοκο, αμφιλεγόμενο και κέρια σημασία ζήτημα. Ελπίζω αμελητή να υπερπηδήσει αυτό το εμπόδιο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύντομα να μπορέσουμε να διαβουλευτούμε με την Επιτροπή για αυτό το ζήτημα, διότι δεν μπορεί η Επιτροπή να απόσχει από τις συζητήσεις που γίνονται στις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές, ε, αυτό όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, αλλά για όλα. Σπάνια συμβαίνει αυτό εξάλλου, οπότε ε, ε, εκπλήσωμαι ακόμη περισσότερο, διότι σας είπα το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, το είπα και το ξαναλέω, είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κινητοποιηθεί και να τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Την Τετάρτη, όπως σας είπα, θα συσκεφθούν οι σκιώδεις εισηγητές. Ελπίζω από αυτή τη σύσκεψη να προκύψουν ενδιαφέρουσες και σημαντικές συμβαστικές λύσεις με τις οποίες θα μπορέσουμε όλοι να ταυτιστούμε και να υποστηρίξουμε. οι σκιώδεις δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε αυτή τη σύσκεψη, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή μαζί μου, με τρόπο ώστε διμερώς να βρούμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στις 18 ε, Σεπτεμβρίου και η Ολομέλεια ε, θα ε, εξετάσει την έκθεση στη, στο δεύτερο Στρασβούργο του Οκτωβρίου. Ο, τώρα κατάλαβα ότι πρέπει να πάω δύο φορές στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο. Ας αφήσουμε το σημείο 10 και ας περάσουμε στο σημείο 11. Eh, έχουμε περιέλθει σε αυτή την, πούς να τη χαρακτηρίσω, λίγο περίεργη κατάσταση όπου απουσιάζει ο επόμενος ηγητής και ο αντικαταστάτης του. Ε, δεν έχουμε εισηγητή εξάλλου για όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις. Οπότε Πρώτη να διακόψουμε για ένα τεταρτάκι. Στις πέντε στις πέντε θα συνεχίσουμε. Ja, okej. Okay. Då så återupptar vi förhandlingarna och utskottsmötet. Συνεχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας. Δηλαδή πήγε 5 η ώρα. Λοιπόν, σημεία 11. Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στον τομέα της ε, ανάπτυξης και της ενισχύσης του κράτους στο Νότιο Σουδάν. Είναι μια γνωμοδότηση που έχει αναλάβει η κυρία Σέσκοβα δεν μπορεί να παρευρεθεί δυστυχώς. Έχουμε τον Καρλ Κόψ που θα μας διαβάσει την παρέμβαση... Α, ο κύριος Κίρκοπ ε, διορθώνει ο πρόεδρος, που θα μας διαβάσει την παρέμβαση κυρία Σέσκοβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη συναδέλφου μου, κυρία Τσέσκοβα, η οποία δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ, όπω πληροφορηθήκατε. Έχει οικογενειακέ υποχρεώσει. Όπω ξέρετε, τα σχολεία αρχίζουν, Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεται εδώ. Ελπίζω να έχετε κατανόηση. Μου ζήτησε λοιπόν να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της έκθεσης και υπάρχουν τρεις ε, τομείς στους οποίους ήθελα να τονίσει σχετικά με τη γνωμοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν θα το πράξω εκ μέρους της. Καταρχάς, στον τομέα της υγείας των ε, μητερών, έπειτα οικογενειακή, ενδοοικογενειακή βία και πρόσβαση σε εξετάσεις για HIV και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Κύριε Πρόεδρε, οι γυναίκε στο Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζουν το υψηλότερο ποσοστό μητρική θνησιμότητα στον κόσμο. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Το να φέρει κάποιο ένα παιδί στον κόσμο στο Νότιο Σουδάν είναι σπάνια ένα χαρμόσυνο γεγονός. Πολύ συχνά οι γεννήσεις οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας είτε της μητέρας είτε του παιδιού είτε και των δύο. Και αυτό είναι κάτι που η συνάδελφός μου θα ήθελε να τονίσει ιδιαίτερα στη γνωμοδότησή της, όπως και έπραξε. Επίσης, το ζήτημα του εξαναγκαστικού γάμου σε μικρή ηλικία και της ενδογενειακής βίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει εδώ εκτενέστατα στην Επιτροπή. Η κυρία Τσέσκοβα λοιπόν θα ήθελε να διασφαλίσει ότι θα αναφερθεί και θα τονιστεί αυτό στη γνωμοδότηση, ιδιαίτερα θα ήθελε να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στις αρχές του Νότιου Σουδάν. Ότι δηλαδή εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουμε την πρακτική και την ανοχή της βίας ενάντια των γυναικών. Οι γυναίκες αυτές εξαναγκάζονται να έρθουν σε γάμο και αυτό πιστεύω είναι κάτι αποτρόπαιο για τους περισσότερους από εμάς. Και η συγγήτρια πιστεύει, πιστεύει ότι η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει λοιπόν να τονιστεί. Επίσης θα ήθελε να αναφερθεί η σημασία της ε, πρόληψης και της υγειονομικής περίθαλψης για το HIV και το AIDS διότι πιστεύει ότι το Νότιο Σουδάν έχει μεν κάνει πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καλωσορίσουμε. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει πολλή δρόμος ακόμα μέχρι οι γυναίκες να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίες υγείας, τις οποίες χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ήθελε επίσης να τονίσει ότι Θα χαρεί πολύ να καλωσορίσετε τα σχόλιά της. Επίσης, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής για τροπολογία σχετικά με τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ποιος θέλει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα, μια που είμαι σκιώδης. Έτσι λοιπόν, όπως ε, είπατε και εσείς, η κυρία Τσέσκοβα δεν μπορούσε να είναι εδώ, αλλά εγώ ως σκιώδης ηγητής θέλω να την ευχαριστήσω και να τη συγχαρώ για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης που μας ετοίμασε. Υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία που αναφέρονται στην γνωμοδότησή της. Αναφέρεται στη βία σε βάρος των γυναικών, το αναφέρατε κι εσείς. Αναφέρεται επίσης ε, στους γάμους των παιδιών. Την παράγραφο 3 άμα μας λέει η κυρία Ανδρέα Σέσκοβα ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις μορφές βίας αλλά και ειδικότερα να αναφερθούμε σε ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νότιο Σουδάν για τον ε, εξαναγκαστικό γάμο. Ε, στο άρθρο, ε, στο σημείο 4, μιλάμε για τη σημασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και τη σημασία που έχουν για την εύρυθμη λειτουργία της ε, κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ε, εργαλείο για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων και την καταπολέμηση της φτώχεια. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την κυρία ε, Τσέσκοβα για την συμβολή της και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρία. Σα ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι τώρα, κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις προτάσεις αυτές που αναφέρονται στην ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και την προστασία των γυναικών στο κράτος του Νότιου Σουδάν. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν δύο προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από εμάς στο Σουδάν. Το ένα έχει να κάνει με τη βία σε βάρος των γυναικών, την αυτονομία και την πρόσβαση στα δικαιώματα των γυναικών και το δεύτερο έχει να κάνει με τον εκδημοκρατισμό μέσω της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των γυναικών. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία έχει ξεκινήσει με δύο προγράμματα τον Ιούνιο και Υπενθυμίζω ότι η αντιπροσωπεία βέβαια για το Νότιο Σουδάν έχει μόλις ξεκινήσει, οπότε ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερα προγράμματα στο μέλλον. Πάντως γενικότερα μιλώντας θέλω να υπενθυμίσω ότι η ΔΕΦΚΟ θεωρεί ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα εγκάσιο θέμα και γι' αυτό και εκπονεί πολλές προσπάθειες και έχει διάφορα μέσα για να ενισχύσει το κράτος δικαίου. Αυτό το κάνουμε μέσω θεματικών εργαλείων για να βοηθήσουμε επιτόπου, αλλά μέσω και κατάρτισης. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο προς αυτή την κατεύθυνση για να διατηρηθεί ισότητα μεταξύ των δύο φίλων σε όλες μας τις δράσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο. Δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Κίχοπ ε, θέλει να πάρει το λόγο και πάλι, όχι έτσι. Όχι, όχι πρόεδρε, θέλω να τονίσω και πάλι πως ε, πιστεύω ότι είναι ύψης της σημασίας το ζήτημα. Δεν έχουμε αθρώα προσέλευση σήμερα το απόγευμα, θέλω όμως να τονίσω ότι η συνάδελφος Τσέσκοβα ελπίζει να αντιληφθούν όλη τη σημασία του ζητήματος και να συμβάλλουν στη δουλειά της. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. 5 ε, Σεπτεμβρίου στι στις 12 είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 3 ε, Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει η ΝΤΕΒΕ για την ίδια έκθεση. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12, σχεδίο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία 2012-2020, καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα. Η συγγήτρια, η κυρία Ρονσούλη, θα πάρει ε, πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή μας ζητήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και όσον αφορά τις τεχνολογίες ICT επικοινωνιών και πληροφοριών. Όταν αυτές εφαρμόζονται κατάλληλα στον τομέα της ε, υγείας, βελτιώνουν την ε, υγειονομική περίθαλψη, το προστόκιμο ζωής και πολλά άλλα. Καταρχάς το σχέδιο δράσης εγκρίθηκε το 2004 και από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει πολλές πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η υγειονομική περιθάλψη στην Ευρώπη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτό, συμμετέχοντας σε πολλά πιλωτικά προγράμματα. Το 2011 η οδηγία για τα διασυνοριακά δικαιώματα των ασθενών και ιδιαίτερα το άρθρο 14 που αναφέρεται στο δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας στοχεύουν στην διασφάλιση περισσότερων οικονομικών και κοινωνικών ε, ωφελών στον τομέα της υγείας. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα ορισμένοι σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσουμε αν θέλουμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για τα διαλειτουργικά αυτά συστήματα. Οφέλη για τους ασθενείς, για τους χειριστές των συστημάτων, για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και για τις αρχές. Η ηλεκτρονική η υγεία μπορεί πολλές φορές να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες που εστιάζουν στον ασθενή και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα ωφέλη και οικονομία χρόνου. Οικονομία χρόνου και μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν και εξοικονόμηση πόρων. Καταρχάς, η έλλειψη πληροφόρησης και εμπιστοσύνης των ασθενών στους επαγγελματίες υγείας, τα μειωμένα ωφέλη κόστους όφελους, η έλλειψη κανόνων και διαφάνειας όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και το υψηλό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας των ε, υπηρεσιών είναι αρνητικά. Υπάρχουν όμως και πολλά ωφέλη και τα ωφέλη αυτά θα τα βρείτε στο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία από το 2012 έως το 2020. Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλές λύσεις και υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το μέλλον, ιδιαίτερα για τις χρόνιες ασθένειες και την ε, αποτελεσματική πρόληψη και προώθηση της. Επίσης, προώθηση της καινοτομίας, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και βελτίωση της ανάληψης ευθύνης Επίσης σημαντικές αρχές είναι η διαφάνεια και η αλληλεγγύη καθώς και η βελτίωση των συνθήκων της αγοράς για την δημιουργία και σωστή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Η γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις σε αυτή μεταξύ των οποίων η πρόταση για διασφάλιση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, για διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στον νέο αυτό τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, η μείωση του κόστους των τεχνολογιών πληροφόρηση και επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο, και επίσης η βελτίωση της κατάρτισης, τεχνικής των γυναικών στον τομέα αυτών, καθώ και η άρση των εμποδίων όσον αφορά την ε, λειτουργική κινητικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η Επιτροπή, ε, ο κύριος Αμπελούς ε, θέλει το λόγο. Ναι, ναι, από τη γάμα Δέλτα Connect. Εδώ υπάρχει το πρόγραμμα δράσης για την υγεία και θα λάβουμε υπόψη μας όσο γίνεται περισσότερο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις προτάσεις σας. Τα συστήματα υγείας, όπως γνωρίζετε, είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αλλά φυσικά δουλεύουμε στα πλαίσια του ηλεκτρονικού δικτύου υγείας με τις χώρες μέλη για να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες που έχουν κάνουν, να κάνουν με την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εδώ αναφέρονται προτάσεις που έχουν να κάνουν γενικά προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό είναι ένα γενικό πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο για τις γυναίκες, για τους ασθενείς, αλλά γενικότερα θέλουμε οι ασθενείς όντω να μπορούν να έχουν πρόσβαση ψηφιακά στα ιατρικά τους δεδομένα, άρα χρειάζεται κάποια κατάρτιση εκεί. Έπειτα για τους παρόχους φροντίδας. Και εδώ πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, να λάβουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουμε την εξάπλωση των δικτύων υγείας. Επικεντρωνόμαστε στους νοσοκόμους για να χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, νοσοκόμες και νοσοκόμοι. Άρα και εδώ θα υπάρξουν τρόποι για να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση ακόμα και οι γυναίκες και οι νοσοκόμοι και οι γιατροί. Προσπαθούμε επίσης να ενσωματώσουμε και τα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας και γενικότερα και για αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική υγεία. Για το κόστος τώρα και τα δίκτυα υπάρχει το κόστος αυτό καθεαυτό το ιατρικό για την τηλεϊατρική για παράδειγμα. Στόχος πάντως του προγράμματος δράσης είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και άρα όσο περνάει ο καιρός να μειωθεί το κόστος των προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας. Υπέρ μεταξύ άλλων και των γυναικών. Όσον αφορά τώρα τις ευκαιρίες για απασχόληση, όντως δεν υπάρχουν ε, αρκετοί άνθρωποι που να έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να απασχοληθούν σε αυτά τα δίκτυα ηλεκτρονικής υγείας. Οπότε ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να φροντίσουν να αποκτήσουν την κατάρτιση αυτή που χρειάζεται για να έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν εκεί. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή των πολιτικών. Οπότε καλό θα ήταν να μπορούμε να παρακολουθήσουμε από πιο κοντά για να δούμε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση, τον ψηφιακό αλφαβητισμό που λέγαμε πριν. Και αν δούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Ρονσούλη, θέλετε το λόγο. Ναι, να προσθέσω δύο πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η υγεία είναι ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Όμως, με στόχο τη μείωση των διοικητικών δαπανών και τη διευκόλυνση της διαχείρισης του συστήματος, ε, πρέπει να αποσκοπούμε προς την ψηφιακή, την ηλεκτρονική υγεία, είναι πολύ μεγάλο το αναπτυξιακό δυναμικό αυτών των ε, τομέων. Ε, ε, να προσθέσω κάποια πράγματα εφόσον έχουμε χρόνο. Ε, το 2012 7,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο δαπανούν τα κράτη-μέλη ε, και λόγω της γέρανας του πληθυσμού και των κοινωνικονομικών κριτηρίων ίσως ε, να αυξηθεί αυτό το ποσοστό και να φτάσει το 8,5% για τις μακροχρόνιες περιπτώσεις περίθαλψης θα διαπλασιαστεί στο μέλλον το κόστος. Οπότε αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο δεδομένα και τα συνδυάζουμε με τις ε, περικοπές ε, στο προσωπικό των νοσηλευτών καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου αυξάνεται ε, υπέρμετρα η αναμονή των ασθενών και νομίζω ότι θα ήταν ωφέλιμες αυτές οι εξελίξεις για όλους όσοι εμπλέκονται στον τομέα της υγείας. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. λίγη συζήτηση. Σήμερα είναι και όπως είπε η κυρία Ρονσούλη, η 5η Σεπτεμβρίου 12 η ώρα το μεσημέρι είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 3 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουν στις 17 Οκτωβρίου και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 13 για τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής προτεραιότητες για το 2013. Η κυρία Κορνέλης, αν έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chair. Um, just... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω λιγάκι το πλαίσιο πρώτα. Πρόκειται για την συνέχεια που δίνουμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε στις αρχές της χρονιάς. Υπάρχουν δύο στιγμές κατά τις οποίες τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, ακούγονται. Με την έκθεση της εικόνων, την Άνοιξη πριν το Ερεινό Συμβούλιο και η δεύτερη στιγμή είναι στα τέλη της χρονιάς, το φθινόπωρο, που πάλι έχουμε έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με γνωμοδοτήσεις από την απασχόληση και τη δικιά μας Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσουμε τι έγινε την χρονιά που πέρασε με το εξάμεινο. Και κοιτάμε βέβαια και τα περί ε, ανάπτυξης και τις προβλέψεις για την επόμενη χρονιά το 2014 λοιπόν. πάντα υπάρχουν πολλά που θέλει κανείς να βάλει σε αυτή την γνωμοδότηση. Οπότε είναι ευπρόσδεκτες και τροπολογίες ώστε αν κάτι έχω ξεχάσει ή αν μπορεί να βελτιωθεί το κείμενο τόσο το καλύτερο. Αυτό λοιπόν εδώ τώρα στη γνωμοδότησή μου που αναφέρω είναι το εξή. Τα κύρια προβλήματα από πλευρά ισότητα των φύλων όσον αφορά το εξάμεινο παραμένουν. αν συγκρίνει κανείς με πέρυσι δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει πολλά. Δεν ε, γίνεται αξιολόγηση όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων όσο αφορά τις επιπτώσεις της λιτότητας, για παράδειγμα, μετά από τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ορισμένες χώρες ε, μέλη κάνουν αυτή τη διάκριση, προσέχουν την ισότητα των φύλων, αλλά στις περισσότερες τίποτα δεν αναφέρεται σχετικά στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ούτε υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με τους στόχους του 2020. Δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και άρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να πούμε αν υπάρχουν διαφορές ή δεν υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες καλές συστάσεις από που έκανε σε διάφορες χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Για παράδειγμα, βελτίωση της μέρημνας για τα παιδιά, κίνητρα, εναρμόνιση της ηλικία ε, συνταξιοδότησης, η αύξηση της μετοχής των γενικών στην αγορά εργασίας και καταπολέμηση του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας. Τα κράτη-μέλη πάντως δεν έχουν ασχοληθεί όσο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια με αυτό το θέμα. Και έτσι εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ισχυρότερη δράση από αυτού. Στο σημείο 6 αναφέρω την ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των διαφόρων φορέων και την υποστήριξη της χρηματοδότησης για συστηματική συμμετοχή των εθνικών φορέων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ορισμένες χώρες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν κάνει ακροάσεις ή κάτι έχουν οργανώσει τέλος πάντων για να φανεί η ανάληψη δέσμευσής τους. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ετοιμάσει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο με κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη για να δούνε πώς θα ενισχύσουν την ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των διαφορών φορέων εκεί είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει για να εστερνιστούν περισσότερο το ευρωπαϊκό εξάμεινο οι διάφορες χώρες. Προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του χρόνου να ετοιμάσει τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη και να φροντίσει να υπάρχει και μια ετήσια ακρόαση με θέμα την ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των διαφόρων φορέων στον τομέα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Περιμένω σχόλια τώρα από εσά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να, μπορώ να ζητήσω ποιος θέλει το λόγο. Αναμένετε εσεί τα σχόλια των συναδέλφων, αλλά είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ και βλέπετε πόσο λιγοστά είναι τα μέλη τη επιτροπή. Είναι λίγο περίεργο. Αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς γίνανε. Μήπως κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Ναι, δεν είναι Ούτε εσεί. Κυρία Ροντσούλη. Ε, θέλω να μιλήσω εξ ονόματος κυρίας Ματέρα. Που ε, ζητάει συγγνώμη και εκείνη για την απουσία της. η Επιτροπή Γυναικών καλεί την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να λάβει υπόψη όλες ιδιαίτερα στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων κατά την εκπόνηση των μέτρων εξυγίανση του προϋπολογισμού. Τα κράτη-μέλη στα εθνικά προγράμματα εξυγίανσης που έχουν καταρτήσει δεν αναφέρονται στην πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων και ε, στην πρόθεση της απασχόλησης. Ε, για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα, στις επενδύσεις. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν εθνικοί στόχοι για την απασχόληση. Ε, ε, με ιδιαίτερο βάρος ε, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τις γυναίκες που έχουν παιδιά σε χαμηλή ηλικία, ηλικία συγγνώμη, χρειάζεται πολυδιάστατη προσέγγιση, διαβίω κατάρτιση, συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία και τα χάσματα ως προς τους μισθούς και τις συντάξεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών θα καταθέσω τροπολογίες με στόχο την κατάργηση ή τουλάχιστον την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Η στρατηγική 2020 ε, προβλέπει 75% ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ε, για τις ηλικίες 20 έως τα 64 μεγαλύτερη συμμετοχή ε, για τους νέους, για τους λιγότερο ειδικευμένους, για τους πιο ηλικιωμένους. Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διακρίσεις που υφίσταται το ασθενές φύλλο στην αγορά εργασίας, στι απαράδεκτε ε, στις απαράδεκτες εργασιακές ε, συνθήκες, τα μισθολογικά χάσματα, την έλλειψη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τα στερεότυπα, τις διακρίσεις που βασίζονται στα φύλλα, αυτά είναι τα βασικά προσκόμματα ε, για την επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στη συνέχεια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο του drop-out, δηλαδή πρόορη εγκατάλειψη της φίτησης ε, που πλήττει κυρίως ε, τα κορίτσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις νέες γυναίκες. Ε, θα καταθέσω τροπολογίες με στόχο τη ρύθμιση αυτών των προβλημάτων. Λαμβάνοντα υπόψη αυτές τις δυσκολίες και εφόσον ε, οι κοινωνικοί κίνδυνοι απειλούν περισσότερο τις νέες γυναίκες παρά τους νέους άντρες, ε, χρειάζεται στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κορνέλης, αν θέλετε μήπως κανά το λόγο για τελικέ παρατηρήσεις. Πολύ σύντομα. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Ροντσούλη αντικατέστησε την κυρία Ματέρα. Πιστεύω πως έφτιαξε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα που με χαρά μου θα συμπεριλάβω στη γνωμοδότηση. Αν υπομονώ λοιπόν να δω τις τροπολογίες. Λυπάμαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας από τους φορείς που αναφέρονται έντονα στην γνωμοδότηση, που κάνουν τόσο πολλά πράγματα για να βελτιώσουν το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν ήταν εδώ για να σχολιάσουν τη γνωμοδότηση. Είμαι σίγουρη όμω ότι θα έχω στο μέλλον την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί του. Ε, Ευχαριστούμε. Εφόσον κανεί άλλο δεν ζητάει το λόγο, ας ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα. 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6. Αυτή είναι η προθεσμή για τις τροπολογίες. 18 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή ε, και στις 30 θα ψηφίσει η ΕΜΒΗ. Πάμε στο σημείο 14. Τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η κυρία αν είναι πάλι εισηγήτρια, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μάλιστα. Πάλι εγώ. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε αυτή τη νέα νομοθεσία, διότι το ζήτημα της διάκρισης των εργαζομένων που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που αυξάνεται Αυξάνεται και επίσης η πίεση από τις πιο λαϊκιστικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στη δική μου χώρα, στην Ολλανδία. Υπάρχουν αρκετά κόμματα, όχι μόνο στα άκρα του πολιτικού φάσματος, αλλά και μεγάλα κόμματα τα οποία δημιουργούν μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα για τους εργαζομένους αυτούς. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ βρίσκεται σε πολύ σωστό δρόμο αναφέροντας ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων θα καταπολεμηθεί μόνο με ε, παρέχοντας ίσα δικαιώματα στους ε, εργαζόμενους που κυκλοφορούν ελεύθερα. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους όσον αφορά τους ε, τομείς τους οποίους ε, δραστηριοποιούνται και στη φύση των διακρίσεων στις οποίες υπόκεινται. Έχω υποβάλει αρκετές ε, προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι αυτοί και ιδιαίτερα οι γυναίκες να είναι καλύτερα πληροφορημένοι για τα δικαιώματά τους. Διότι εκεί είναι και η αφετηρία. Οι άνθρωποι που ζητούν να πληροφορηθούν για τα δικαιώματά τους πρέπει να έχουν το δικαίωμα λοιπόν και να πληροφορούνται και να μπορούν να τα ασκήσουν. Ιδιαίτερα οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν τι πληροφορίες υπάρχουν όσον αφορά τη στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, την οικογενειακή κατάσταση, επιδόματα για την ε, παιδική μέρη άδεια μητρότητας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε την αυτοργάνωση των εργαζομένων αυτών. Αυτό πιστεύω θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς είναι προς το συμφέρον τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους και τους οικιακούς βοηθούς, οι οποίοι πολλές φορές έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά αυτοργάνωσης και γίνονται θύματα διακρίσεων περισσότερο από ότι οι εργαζόμενοι σε άλλους τομείς. Επίσης, χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην διάσταση του φύλου και στο γεγονός ότι πολλοί από τους εργαζόμενους αυτούς ε, φέρνουν και τις οικογένειές τους μαζί στις χώρες τις οποίες ε, εργάζονται. Επίσης, ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι η αναγνώριση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών ή των συμφώνων συμβίωσης. Είναι μια επιλογή που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, το να μην δηλαδή έρθουν σε γάμο, αλλά το να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο. Και αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται διασυνοριακά, καθώς επίσης και τα σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους. Ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή να στηρίξει τη γνωμοδότηση αυτή και να προσθέσει ό,τι χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Κυρία Ρονσούλη. Ναι, ναι, εδώ είμαι κι εγώ. Ακόμα. Τώρα πάλι θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Ματέρα. Ένας από τους κύριους πυλώνες για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, που πρέπει να βασίζεται στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ρύθμιση του 2011, το άρθρο 45, δίνει στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διάκριση εξαιτία της επικότητάς τους. Παρ' όλα αυτά παραμένουν διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που μετακινούνται από μία χώρα στην άλλη και βασίζεται αυτή στο φύλλο πολλές φορές, στην προέλευση, την καταγωγή, τη θρησκεία. Οι τροπολογίες της κυρίας Κορνέλισον με βρίσκουν σύμφωνοι σε ένα μεγάλο βαθμό. Η τροπολογία 1 με βρίσκει σύμφωνη γιατί υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Συγχρόνως σέβεται την αρχή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και της ίσης μεταχείρισης ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνώ όμω εξίσου με τις τροπολογίες 4 και 5, γιατί στις τροπολογίες αυτές γίνεται μνήα στην ε, ε, συμβίωση των ε, σεξουαλικό προσανατολισμό, κάτι το οποίο νομίζω ότι ξεπερνάει το θέμα της Επιτροπής Γυναικών. Όσον αφορά την τροπολογία 6, δεν συμφωνώ με όλο το θέμα των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Το τελευταίο μου σημείο είναι εκείνο που λέει ότι πρέπει την τροπολογία αυτή να την εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και να φροντίσουν για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες μεταξύ και γυναικών στον τομέα της αγοράς εργασίας. Με αυτό συμφωνώ. Είναι αναγκαίο. Πάντω, το άρθρο 5 θα προσπαθήσω να το τροποποιήσω περισσότερο. Η τροπολογία της κυρία Κορνέλσον πιστεύω ότι δεν πηγαίνει αρκετά μακριά. Πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα τη διάκριση εξαιτία του φύλου και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε οργανώσεις που θα ασχοληθούν για να πετύχουν το στόχο αυτό. Είμαι κατά των τροπολογιών 19 και 20 γιατί νομίζω ότι δεν εμπίπτουν στο θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής Γυναικών δηλαδή. Τροπολογία 28 τώρα. Αυτή νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι σαφές εδώ για το ποια συμφέροντα υποστηρίζονται. Καλώς. Δίνω τώρα το λόγο. Α, παρακαλώ κυρία Μπάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι στην Επιτροπή Απασχόλησης η συγκίτρια για αυτό το θέμα. Έχουμε υπόψη μας ότι η κατάσταση είναι τέτοια που από όλες τις ελευθερίες, η ελευθερία διακίνησης είναι αυτή που χρησιμοποιείται λιγότερο. Και αν συγκρίνουμε τα δύο φύλλα, διαπιστώνουμε ότι η αναλογία γυναικών είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη των ε, ανδρών που κυκλοφορούν δηλαδή για να εργαστούν ε, σε άλλη χώρα από τη δικιά τους. Στην έκθεση αυτή λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε για μετανάστες, για μετανάστευση. Εδώ μιλάμε για την κινητικότητα των εργαζομένων. Γι' αυτό και αλλάζουμε και την ορολογία. Το θέμα της συλλογικής αποζημίωσης είναι επίσης κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποτελεί νομοθεσία. Θέλουμε να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν, να ενισχύσουν, να εφαρμόσουν τη δυνατότητα οργανώσεων που θα εκπροσωπούν τους εργαζόμενους από την πρακτική η δικαστική αποκατάσταση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε ποια οργάνωση μπορεί να βοηθήσει. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σημείο επαφής και να υπάρχει και ένα δίκτυο τέτοιων σημείων επαφής. Γιατί σε αυτή την γνωμοδότηση έχει μεγάλη σημασία και το θέμα της ερμηνείας συγγνώμη, το κόστος της μετάφρασης σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος της μετάφρασης των ε, γράφων που μερικές φορές είναι εκατοντάδες και εκατοντάδες. Στο σχέδιο της Επιτροπής, διότι πολλές φορές σελίδε ε, από το Solvit που έχουν να κάνουν αυτό το θέμα είναι πολλές. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να καλύψουμε το θέμα με τέτοιο τρόπο που να είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να οργανώσουν μια τέτοια δομή, αλλά να βρούμε και ποιος στην κάθε χώρα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για τα διάφορα ζητήματα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ πολύ με την προσέγγιση που ακολουθεί η γνωμοδότηση αυτή και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι γυναίκες πολύ πιο δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ελευθερία αυτή γιατί ζουν σε πιο περίπλοκες καταστάσεις μια που εκείνες καλούνται να συμφιλιώσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα άρθρα η διάσταση του φύλου, αλλά αυτό που είναι ίσως δυνατόν είναι να διευρύνουμε το εύρος της νομοθεσίας αυτής. Γιατί όπως γνωρίζουμε έχουμε και άλλες νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με την διάκριση των δύο φύλων. Είναι αδύνατο λοιπόν να συμπεριλάβουμε όλα τα προβλήματα. Πώς να διασφαλίσουμε την μη διάκριση σε βάρος ορισμένων πολιτών από άλλη χώρα. Άλλο θέμα είναι οι δικαστικές ε, υποθέσεις. Αν περιορίσουμε τα ευρωσεφαρμογής, γιατί το άρθρο 45 τελειώνει με τη διατύπωση που λέει ότι η ελευθερία περιορίζεται σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις Οι δικαστικές αποφάσεις όμως διαφέρουν. λένε ότι υπάρχει περιορισμός σε ορισμένα επαγγέλματα για ορισμένους πολίτες οι οποίοι έχουν να κάνουν με εκτελεστικές δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή είναι μια γνώση που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας στη γνωμοδότηση αυτή. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες προτάσεις που όντως ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογή της ρύθμισης αυτής. Τροπολογίες που έχουν να κάνουν με άλλες οδηγίες κατά των διακρίσεων. και όχι αυτές που περιορίζονται στους Ευρωπαίους πολίτες. Εν κατακλείδη. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που έκανε η συγκήτρια. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά έκανα ό,τι μπορούσα για να επικεντρωθώ στη διάσταση του φίλου και να λάβω υπόψη μου τις προτάσεις εκείνες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης αυτής. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, πολύ σας ευχαριστούμε. Έχουμε και τον κύριο Πιέρης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι ε, πολύ σύντομος. Καλώς ορίζουμε λοιπόν το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Δύο σημεία θα θέλαμε να θίξουμε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση αυτή δεν στοχεύει στην ε, επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 492. Ούτε δηλαδή να το επεκτείνει, ούτε να το περιορίσει. Θα θέλαμε λοιπόν να σας παραπέμψουμε στην πρόταση υδροπολογίας 3, όπου γίνεται αναφορά στην Οδηγία 2004-38 Εκεί το πρόβλημα που παρατηρούμε είναι ότι η οδηγία 2004-38 δεν καλύπτει τους εργαζομένους σε, στα σύνορα. Μία προστίκη λοιπόν θα δημιουργήσει σύγχυση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οικογένειες των εργαζόμενων στις ε, παραμεθόριες περιοχές, στις μεθοριακές περιοχές, με συγχωρείτε. Να σας επιστήσουμε λοιπόν την προσοχή σε αυτόν τον κίνδυνο. Έπειτα, οι τροπολογίες 12 έως 16. οι οποίες αφορούν και αυτές το πεδίο εφαρμογή, κάποιες λεπτομέρειες σχετικές με αυτό. Θεωρούμε πως όλες αυτές, αν όχι οι περισσότερες από αυτές, καλύπτονται ήδη από την διατύπωση του κανονισμού 492. Η ερμηνεία του δικαστηρίου για το κοινωνικό πλεονέκτημα είναι αρκετά ευρία. Ορισμένες ε, τροπολογίες λοιπόν από αυτές ενδεχομένως να καλυφθούν από την απόφαση του δικαστηρίου. Μία πιο συγκεκριμένη αναφορά από αυτές τις τροπολογίες ενδεχομένως περιορίσει την έννοια του κοινωνικού πλεονεκτήματος. Θα θέλαμε λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Αυτά λοιπόν για το κοινωνικό πλεονέκτημα και τώρα όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης. Και αυτό ένα ευρύτατο θέμα. Και εδώ καλύπτονται αυτά αυτές οι τροπολογίες από σημεία που ήδη υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και τροφαρμακευτικής περίθαλψης, αυτά καλύπτονται από τον κανονισμό 883 για την κοινωνική ασφάλιση. Θεωρούμε λοιπόν ότι και εδώ δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μνήα στα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στην οδηγία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρία Κορνέλισεν, έχετε τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και τους τρεις. Η κίνδυνη που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλό να το κοιτάξουμε ιδιαίτερα, διότι φυσικά δεν είναι αυτέ οι προθέσει μου, να αποκλείσω δηλαδή ορισμένες ομάδε εργαζομένων ή να περιορίσω τα κοινωνικά πλεονεκτήματα. Το αντίθετο επιθυμώ. Θα χαρώ λοιπόν πολύ να συνομιλήσουμε ξεχωριστά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Κύρια Ματέρα, χαίρομαι πολύ που στηρίζετε ορισμένες τροπολογίες και εκείνες που δεν τις στηρίζετε είναι κάτι που δεν με εκπλήσει. Θα χαρώ λοιπόν να συζητήσω μαζί σας περαιτέρω. Κύριε Μπάουερ, αναφέρατε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, ότι δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με το ποιος ευθύνεται και ποιος όχι. Αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε. Τώρα, πέρα από το πεδίο εφαρμογή, δεν έχω πρόβλημα να επεκταθώ πέραν του πεδίου εφαρμογής εάν αυτό είναι δυνατόν και αν δεν αποτελεί μειονέκτημα. Απομένει να δούμε πόσο μπορούμε λοιπόν να τεντώσουμε τα όρια του πεδίου εφαρμογή. έτσι ώστε να βελτιώσουμε την οδηγία και να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους μετακινούμενους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε αρκετά ευάλωτη θέση, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Και να προσπαθήσουμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα κλείνοντας να σας πω ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες είναι πάλι 5η Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, 5 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 3 Οκτωβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή μας και στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, τώρα κλείσαμε και το σημείο 14, το επόμενο σημείο είναι η προσεχή συνεδρίαση 18 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και την ίδια μέρα από τις 3 μέχρι τις 6.30. Σας ευχαριστώ λοιπόν για σήμερα και καλό βράδυ σε όλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE